Μια διαδικαστική πρόταση. Ζητούμε ένα νέο σημείο, μια ερώτηση προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα μάθαμε ότι οι αρχές της Νορβηγίας τελικά απέσυραν ένα παιδί από την ε, μητέρα του και το έδωσαν σε μια οικογένεια υποδοχής. Είναι απαράδεκτο αυτό. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε και να κάνουμε τίποτα για να προστατεύσουμε τα παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ζητώ, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, να στηρίξετε την ερώτησή μας και να μπει αυτή στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Έχετε δίκιο, κυρία μου. Όμως, πρέπει να περάσετε από την συνδιάσκεψη των Προέδρων. Αν θέλετε να εγγραφεί το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, θα το κάνουμε. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης, υπάρχουν σχόλια ή παρατηρήσεις. Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης. Και θα περάσουμε στην προφορική ερώτηση.